πληρώσουν την κρίση εκείνοι οι οποίοι ευθύνονται για την κρίση. Αυτό που χρειάζεται τώρα δεν είναι περικοπές ε, προς πάσα κατεύθυνση. Θα πρέπει ε, να βοηθηθούν οι χώρες... Α, ο πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή, τελείωσε ο χρόνος. Ευχαριστώ. Ο Mr. please. Ο κύριος Πετρουλούχαν. Ευχαριστώ, πρόεδρε.